Περνάμε στι επεξηγήσει ψήφου και ξεκινάμε με την έκθεση Νταζάν για την εφαρμογή της κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνα. Δίνω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Χάναν. Κύριε Χάναν. Κύριε Χάναν, Ντάνιελ Χάναν, έχετε το λόγο. Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τι περίεργη ιδέα την ε, εξωτερική πολιτική να την ε, διεξάγουμε από κοινού. Να μην μπορούμε να επηρεάσουμε τον κόσμο ως ανεξάρτητες φωνές. Δείτε το παράδειγμα της Νορβηγίας που δεν ανήκει στην ε, Ένωση. 9 εκατομμύρια διπλωμάτες της χώρας αυτής όμως δραστηριοποιούνται σχεδόν ε, σε όλες τις υπήρους και αρχιπέλαγα ε, την Ειρηνευτική Συμφωνία μεταξύ Σουδάνου Του Σουδάν, συμφωνία του Όσλο μεταξύ Παλαιστίνης Ισραήλ, στη Σρι Δραστηριοποιούνται σε όλες αυτές τις συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Μια μεγάλη χώρα μπορεί επομένως να επηρεάσει και τις παγκόσμιες υποθέσεις. Το Ενωμένο Βασίλειο, 63 εκατομμύρια την ναυτική χώρα, εμπορική χώρα ε, και ε, διανόμου και παραδόσεως είχε σχέσεις εμπορικές με όλες τις υπήρους. Ως πέμπτη παγκόσμια οικονομία και τέταρτη στρατιωτική δύναμη στάτους δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα είδος ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής ε, διακόπτη πρόεδρος. Για ένα λεπτό κυρία Γκίλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ενώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα επιταχύνουμε τη συνεργασία για την ΚΕΠΑ και για να γίνει πιο αποτελεσματική, έχει σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, να συμμετάσχει. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία, αλλά αν υπάρχει επικάλυψη ως προς ε, ε, δράσεις του ΝΑΤΟ, δεν έχει νόημα να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι κατασπαταλούμε το δημόσιο χρήμα. Νομίζω όμως ότι η έκθεση ασχολείται με θέματα ύψης της σημασίας που θα πρέπει να μας απασχολήσουν τη στιγμή που θα συζητήσουμε την ΚΕΠΑ τον Ιούνιο. Θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία με τους ελάχιστους ε, πόρους που διαθέτουμε. Διακόπτη Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πολτσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι η ΚΕΠΑ είναι κάτι το πολύ σημαντικό η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Θα πρέπει να είναι μια ενιαία πολιτική γιατί θα ήμασταν πιο ισχυροί και θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ισχυρότερη φωνή στη παγκόσμια σκακέρα. Και σε σχέση με την πολιτική άμυνας, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη με τον ΝΑΤΟ. Φυσικά δεν πρέπει να υπάρχουν ε, ε, επικαλύψεις από εμάς των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ, αλλά η κατάσταση στην Ουκρανία δείχνει ότι χρειαζόμαστε μία σαφή λύση. Κύριε Ζιάρ. Για μας, Πρόεδρε, το ζήτημα δεν είναι αν πρέπει ή αν μπορεί να προσφέρει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Πρέπει, οφείλει, πιστεύω, να προσφέρει περισσότερα. Αν κοιτάξουμε στο παγκόσμιο σκηνικό τι συμβαίνει έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να διαρωτηθούμε εάν έχει καταστεί πιο σταθερή η κατάσταση ή όχι. Και μάλλον έχει συμβεί το δεύτερο. Άρα χρειάζεται μια περισσότερη προσπάθεια στην πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Υποστηρίζουμε λοιπόν την έκθεση. Θα ήθελα μόνο στις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προκύψει ένα, αποτέλεσμα, ένα πόρισμα. Δεν μπορούμε να έχουμε διπλές δομές. Πρέπει τα κράτη-μέλη μαζί ε, με, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να είναι διαθέσιμα, να είναι διατεθειμένα να θεσπίσουν μια πολιτική ασφάλεια και άμυνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Γούλφ. Ευχαριστώ. Ένα χρόνο πριν ήμουν εδώ στο σώμα ως νέο μέλος. Όταν έγινε λόγος για κυρώσεις κατά της Ρωσίας και όταν μιλήσαμε και για πόλεμο κατά της Ρωσίας, τους είπα μην ανησυχείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ε, τέτοιες βλέψεις αλλά με την πολιτική αυτή, μια κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, το σώμα ε, ψήφισε τη χρηματοδότηση ενός στρατιωτικού σώματος, ε, την στρατιωτική έρευνα καθώς και φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις άμυνας καθώς και τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσει ε, μια νέα δραστηριότητα ως προς τα μη επανδρομένα οχήματα. Νομίζω ε, ότι γι' αυτό επιβαλόταν να καταψηφίσω γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προβάλλει πόλεμο κατά άλλων κρατών. Επόμενη έκθεση Κούκαν και Ταράντ, χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η κυρία Γκίλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ξαναδούμε την κοινή μας πολιτική άμυνας και ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους ωφελίας της ΣΚΕΠΑ για να δούμε πώς μπορούμε να επιμερίσουμε τους ε, πόρους και την ικανότητά μας για έχουμε πιο ευέλικτες αποστολές σε ΚΕΠΑ για να προβάλλουμε την εξωτερική μας πολιτική, καλύτερη διαχείριση των πόρων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε συμπληρωματικό χαρακτήρα με αυτά που γίνονται αλλού, όπως το ΝΑΤΟ. Αλλά δεν θεωρώ ότι χρειάζονται φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις εξοπλισμών, γιατί η συνεργασία υφίσταται κάθε αυτή και δεν χρειάζεται φορολογικά μέτρα που θα μείωναν την αποτελεσματικότητα των αποστολών. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι ε, πέντε χρόνια πριν δεν γινόταν ε, λόγος για θέματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά μετά από την κατάσταση στην Ουκρανία και τη συμμετοχή της ε, Ρωσίας στην εμπόλεμη κατάσταση, πολλές χώρες άλλαξαν στάση και αναθεωρούν. Και φαίνεται ότι το ίδιο κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ψήφισα με την ομάδα μου ε, για όλα, εκτός από το άρθρο 3, την παράγραφο 2. Ε, απόσχαμε από αυτό το άρθρο γιατί μιλά για στρατιωτικό χαρακτήρα, στρατιωτικές δράσεις και στην Ιρλανδία θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι όπως είμαστε και σε όλα τα άλλα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Εάν δεν βλέπω κάποιον που έχω στη λίστα μου, στην αίθουσα δεν θα τον καλώ. Περνάμε στην έκθεση Γκόμες, δυνατότητες ασφάλειας και άμυνα στην Ευρώπη. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκίλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απήχα στην ψηφοφορία τη εκθέσεω, διότι είμαι, είμαι, είμαι λίγο επιφυλακτική σε αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτή, για αυτή την πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Ε, είναι οι ανησυχίε μου παρόμοιε με αυτέ που εξέφρασα και για άλλε παρόμοιε εκθέσει. Θέλω όμω να τονίσω ότι τίθενται διάφορα κρίσιμα ζητήματα και θα ήθελα να τα αντιμετωπίσουμε εντελεχώ ε, στη συνάντηση του Ιουνίου ε, των Υπουργών Άμυνα και των ηγετών των Αρχαιοκράτων και κυβερνήσεων. Κυβερνοχώρο είναι ένα σημαντικό θέμα. Ε, υπάρχουν απειλές στην ασφαλειά μας. Θεωρείται όμως πολύ συχνά ως απειλή που έχει να κάνει με το μακρινό μέλλον. Όμως ε, είμαστε πολύ πίσω. Ε, δεν χρησιμοποιούμε στρατηγικά τον κυβερνοχώρο για να προσπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας. Στο παγκόσμιο προσκήνιο όμως είπα κάθε χρόνο ορίζει τι κυβερνοεπιθέσει ω την σημαντικότερη απειλή προς την εθνική ασφάλεια. Στην Ευρώπη ούτε καν στο ραντάρ δεν την έχουμε αυτή την απειλή. Επόμενο, ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Αν θέλουμε να φροντίσουμε για την κοινή μας ασφάλεια. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν ε, από κοινού μεταξύ των κρατών μελών. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε μια φωνή στο ΝΑΤΟ. Ε, μια ενιαία φωνή εκεί, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών ε, είναι μέλη αυτού του οργανισμού, αυτού του συμφώνου. Για ποια κοινή πολιτική όμως μπορούμε να μιλάμε όταν 7 χρόνια μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Γεωργίας οι φίλοι μας ε, από τη Γεωργία δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και σε αυτή την επταετία μέσα δεν έχουμε μιλήσει με μία φωνή για την ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, κοινά θεσμικά όργανα, κοινέ αρμοδιότητες, όλα αυτά ε, πρέπει να εφαρμοστούν για ε, να γίνει πιο ισχυρή η κοινή μας πολιτική ασφάλειας και να μην είναι μόνο μια πολιτική που φαινομενικά φαίνεται να είναι επωφελής, αλλά τελικά βλάπτει τα συμφέροντα των κρατών μελών. Πρόεδρος, επόμενη έκθεση θα ήταν η έκθεση πρόοδου του 2014 για την Τουρκία, αφού όμως ψηφίσαμε αναβολή αυτής της εκθέσης και γνωρίζω ότι έχουν καταλήψει την αίθουσα από που ήθελα να λάβουν το λόγο. Ο κύριο Κέλλη ήταν ο μόνος που παρέμεινε. Παρ' όλα αυτά δεν θα έχουμε επεξηγήσει ψήφου για αυτή την έκθεση και εδώ ολοκληρώνουμε τη διαδικασία επεξηγήσεων ψήφου. Θα ε, υποβάλουμε τα πρακτικά στις αρχές επόμενη συνεδρία προ έγκριση και αν δεν υπάρχει ε, κάποια αντίρρηση μαζί με τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν ε, σήμερα. Θα